Αγαπητοί συνάδελφοι, άρχεται η συνεδρίαση. Νομίζω μπορούμε να αρχίσουμε. Καταρχήν, ε, να σας ζητήσουμε συγγνώμη που καθυστερήσαμε λίγο να αρχίσουμε, γιατί είχαμε προτάξει τη συνεδρίαση των συντονιστών και δεν κατορθώσαμε να τελειώσουμε ακριβώς την ώρα μας. Δεύτερον, θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσον συμφωνείτε με την ημερήσια διάταξη. σημείο 3 έχω να κάνω μία ανακοίνωση. Δηλαδή, το σημείο υπαριθμών 13 της ημερήσιας διάταξης ε, διαγράφεται γιατί δεν είναι παρόν ο συνάδελφος. Και επίσης ε, να σας επισημάνω ότι σήμερα το απόγευμα θα ξεκινήσουμε αργότερα γιατί έχει ολομέλεια το μεσημέρι απλά για ενημέρωσή σας. Και επίσης ε, αύριο στην ακρόαση είστε βέβαια προσκεκλημένοι να παραστείτε και αυτή η ακρόαση θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί από τον κύριο Ταγιάννη και τη συζητή στην παρουσίασή του ε, θα έχουμε πολλά ενδιαφέροντα θέματα για τους επόμενους μήνες. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε κατά τη διάρκεια των διακοπών και να μπορούμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Πάμε στο σημείο υπαριθμών 4 και ρωτώ κατά πόσον ε, στα πρακτικά έχετε να κάνετε κάποια παρατήρηση. Από ό,τι βλέπω όχι, ως εκ τούτου εγκρίνονται τα πρακτικά. Πάμε στο σημείο υπαριθμών 5. Πρόκειται για την καινοτομία, πολιτική καινοτομία και θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, στο συνάδελφο κύριο Βίνκλα, ε, Χτες ε, δεν θέλαμε να γίνει συνεδρίες και αναγκαστήκαμε να αναβάλουμε το θέμα αυτό. Κύριε Βίνκλερ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα το αναβάλαμε, αλλά δεν κατορθώσαμε να κερδίσουμε περισσότερο χρόνο. Θα τα πω πάρα πολύ γρήγορα για να προλάβω μέχρι την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Καταρχήν ευχαριστώ όλους ε, τους ε, άμεσα εμπλεκόμενους ε, για τις διμερείς επαφές, αλλά και για τις τροπολογίες που κατέθεσαν. Συνολικά λοιπόν... Έχουμε 108 τροπολογίες, κάτι που για την έκθεση αυτή είναι πολύ ικανοποιητικό ο αριθμός. Βέβαια πρέπει να προσέξουμε για το ότι αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις εξελίξεις ε, κυρίως ε, στην οικονομία και στην κοινωνία. Ως εκ τούτου το θέμα δεν θα πρέπει να επιβαρυνθεί με την ε, προσθήκη πολλών τροπολογιών. Σε τελική ανάλυση, άμα γίνει αυτό, δεν θα μπορεί κανείς να διαβάσει την έκθεση. Προτείνω λοιπόν να απλουστεύσουμε την έκθεση για να γίνει καλύτερα κατανοητή. Και επίσης προτείνω ε, να γίνει κάποια σύντμηση, κάποια κάποιο συντονισμό των ε, τροπολογιών. Υπάρχουν κάποιε τροπολογίε οι οποίε προέκυψαν από την ανταλλαγή απόψεων εδώ στην Επιτροπή, επίση από τι παρεμβάσει συναδέλφων και αυτό που ενδιαφέρει είναι από κοινού α πούμε με τη συνάδελφο κυρία Ντεκαστήλιο τα σημαντικά θέματα όπως είναι ο επιμερισμός ε, κινδύνων ε, στη χρηματοδότηση ή δείκτες ε, καινοτομίας για συνέργειες στα διάφορα προγράμματα πλαίσιο και τα διαρθρωτικά ταμεία ή θέματα που έχουν σχέση με την ομάδα εμπειρογνωμόνων και κυρίως για την τεχνολογία κλειδί τα θέματα της υπεραξίας ή αν θέλετε το σημαντικό θέμα για τον συντονισμό ανάμεσα στις ε, διάφορες ε, γενικές διευθύνσεις. Αυτές είναι σταχυολογώντας ε, κάποιες τροπολογίες που κατέθεσα εγώ και ορισμένοι συνάδελφοι φαντάζομαι θα είναι ικανοποιημένοι. Υπήρξαν συζητήσεις με, παραδείγματος με την κυρία Μέρκης η οποία είναι υπέρ της ε, διαγραφής ε, κάποιων δικών μου τροπολογιών. Βέβαια υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας και εγώ θέλω να πω το εξής. Αυτό που ενδιαφέρει κυρίως είναι όχι μόνο να προάγουμε τα υπάρχοντα όσον αφορά την καινοτομία και τη βιομηχανία, αλλά να προάγουμε και τη δημιουργικότητα να προωθήσουμε το καινούριο έτσι ώστε να υπάρξουν νέες επιχειρήσεις βεβαίως προβλέποντας την απαραίτητη χρηματοδότηση και τη στήριξη των ε, καινοτομιών. Να δώσουμε περιθώριο ελιγμών σε αυτές τις νέες επιχειρήσεις να κινηθούν και στην αγορά και στον ε, χώρο της ε, βιομηχανίας. Επειδή δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας, θα ήθελα να πω κάτι που αφορά στους εκπροσώπους της Κομισιόν που παρίστανται. Να τους πω λοιπόν ότι όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και σε σχέση με την καινοτομία ε, θέλουμε να ξέρουμε κατά πόσον ε, ο τίτλος που υπάρχει θα παραμείνει ή θα επιλεγεί κάποιος άλλος. Παραδείγματος χάρη ε, πρόγραμμα έρευνας για την καινοτομία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό έτσι ώστε οι αρμόδιες γενικές διευθύνσεις να μπορούν να δρομολογήσουν την ικανοποιητική συνεργασία. Να γνωρίζουμε πώς ακριβώς θα δουλέψει η ομάδα κρούσης, ποια θα είναι η συνεργασία και πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα. Αυτά είναι ήδη εισαγωγή και σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, ε, λέει ο Πρόεδρος, και θέλω να δώσω το λόγο πρώτα απ' όλα στη συνάδελφο κυρία Μέρκης. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βίγκλερ για την ε, συνεργασία και την ε, εξαιρετική έκθεση. Θα ήθελα όμως να τονίσω ότι θα πρέπει να προβούμε σε μία διαρθρωτική αλλαγή. Χρειαζόμαστε μία διαφορετική κοινωνία. Βεβαίως καταπολεμούμε τις κλιματικές αλλαγές, αλλά γιατί να μην προωθήσουμε μία βιώσιμη κοινωνία και να μην καταπολεμούμε απλώς και να προβούμε και σε διαρθρωτικές αλλαγές στο μεταξύ. Αυτή η έκθεση τονίζει ότι η κοινοτομία είναι κλειδί για μια βιώσιμη κοινωνία και δεν θα πρέπει να εστιάσουμε μόνο στις οικονομικές απολαβές για τις ε, επιχειρήσεις, κάτι το οποίο είναι σημαντικό, αλλά θα πρέπει να μας ενδιαφέρουν και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ωφέλη. Στην έκθεση καταγράφεται ότι είναι αναγκαίο να μην υπάρχει χάσμα μεταξύ έρευνας, και καινοτομίας και αγοράς διότι χρειαζόμαστε εμπορεύσιμα πράσινα προϊόντα στην καινοτομία. Θα πρέπει λοιπόν να πληρωθεί αυτό το χάσμα. Και αυτό σημαίνει και συμμετοχή των πολιτών διότι η καινοτομία δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη τόνωση και δημιουργικότητα. Άρα για να καινοτομήσουμε χρειαζόμαστε καλύτερη εκπαίδευση, καλύτερο σύστημα ε, όθησης και τόνωσης της ε, καινοτομίας. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε μια οριζόντια και εγκάρσια προσέγγιση, δηλαδή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών, αλλά και μεταξύ θεσμικών οργάνων και μέσα στα θεσμικά όργανα, διότι θα πρέπει να έχουμε μια καλύτερη οριζόντια προσέγγιση εντός Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να εστιάσουμε την προσοχή μας ο καθένας της ε, στην ειδικότητά του για να δούμε ποια θα είναι τα ωφέλη για την καινοτομία. Τέλος, θα πρέπει να δούμε τις πρώτες ύλε το θέμα των πρώτων υλών, διότι χρησιμοποιούμε σπάνιες πρώτες ύλε για την καινοτομία και θα πρέπει να δούμε το, το θέμα της σπάνιδος και της καινοτομίας. Αυτό θα πρέπει να είναι το επίκεντρο των ε, σκέψεων μας, της σκέψης μας. Γι' αυτό θα ήθελα η Επιτροπή να ασχοληθεί και με το θέμα της ε, σπάνιδος των προϊόντων το οποίο ε, χρησιμοποιούμε στην καινοτομία. Σας ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον κύριο Τάκουλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γουίνκλερ για την εξαιρετική αυτή εργασία. Όταν ε, δούμε, όταν βλέπουμε την έκθεση και θυμάμαι και το υπόβαθρο της έκθεσης, θα πρέπει να διατυπώσουμε μια έκθεση και να δώσουμε τα μέσα στην Κομισιόν για να φτάσει σε αυτό το απότερο μέσο. Αν δούμε τους απότερους στόχους και την πρόταση, ε, οι 100 τροπολογίες είναι πολλές. Η παρουσίαση του κυρίου Βίνκλερ θα πρέπει να είναι επαρκής. Θα πρέπει να δούμε την προστιθέμενη αξία των τροπολογιών, αν υπάρχει γιατί θα πρέπει να προωθηθούν καταλήλως. Πολλές φορές ε, δεν σκεφτόμαστε την προστιθέμενη αξία, απλώς θέλουμε εμείς να αφήσουμε το αποτύπωμά μας σε αυτά τα έγγραφα. Δεν θα πρέπει να μας απασχολεί αυτό, θα πρέπει να μας απασχολεί η Ευρώπη και κάτι άλλο. Την προηγούμενη εβδομάδα στην Φιλανδία Ε, μία εφημερίδα ασχολήθηκε με τους πιο επιμελείς ε, βουλευτές και είπε ότι οι πιο επιμελείς είναι αυτοί που υποβάλλουν στις περισσότερες τροπολογίες. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Οι πιο επιμελείς βουλευτές είναι αυτοί που προβάλλουν συμβιβασμούς. Και ο κύριος Βίνκλερ έχει μια πολύ καλή βάση εργασίας, άρα η δική του παρουσίαση θα πρέπει να αρκεί. Άρα όσοι υποβάλλετε τροπολογίες θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε. Προσφέρουν κάτι περισσότερο στην έκθεση, εγώ δεν νομίζω. Δηλαδή, όσοι περισσότερους μάγειρες έχουμε στην κουζίνα, τόσο χειρότερη θα είναι η σούπα. Πώς μπορούμε λοιπόν να φτάσουμε στη, στην ουσία, στην πεμπτουσία αυτής της παρουσίας, αυτής της έκθεσης. Γι' αυτό υποστήριζω τον κύριο Βίνκλερ. Ο κύριος Μπιτικόφα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον ε, κύριο ε, Βίνκλε για την μέχρι τώρα εργασία του σε αυτό το θέμα και τον συγχαίρω όχι μόνο για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το θέμα της ε, καινοτομίας. Στο σημείο αυτό συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε η κυρία Μέρκης, δηλαδή παρουσίασε με θαυμάσιο τρόπο την προσέγγιση που πρέπει να υιοθετήσουμε, δηλαδή η καινοτομία να ερμηνεύεται ως ε, μια ε, κοινωνική διεργασία με την ευρύτερη έννοια ε, της λέξης κοινωνικός. Με τον κύριο Βίνκλερ είχαμε συζητήσεις και βλέπω κάποια στοιχεία που τις συζητήσεις αυτές τα έχει υιοθετήσει. Και εγώ σε αντίθεση με τον προαλήσαντα δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει πρόβλημα με τις τροπολογίες. Οι τροπολογίες μπορούν να υιοθετηθούν γιατί οι τροπολογίες αυτές κατά την άποψή μου έχουν προκύψει μετά από συνεργασία. Θα ήθελα να επισημάνω κάποια σημεία τα οποία ενδιαφέρουν εμένα και νομίζω ότι ε, υιοθετώντα τα σημεία αυτά μπορούμε να βελτιώσουμε την έκθεση. Πρόκειται πρώτα απ' όλα για την προβολή του ρόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο θέμα της καινοτομίας. Κατά δεύτερον, θεωρώ ότι πρέπει να προβάλλουμε περισσότερο τις ε, οικολογικές καινοτομίες. Και εδώ τίθεται το θέμα της επάρκειας ε, των πόρων, κάτι που έδειξε και η κυρία Μέρκες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κατόπιν, πρόκειται για τα κλάστες, για, τα, για τους περίφημους ε, συνεργατικούς σχηματισμούς γνώσης. Και το τελευταίο θέμα αυτό θέλω να σας το πω και εγώ, γιατί έχουμε καταθέσει εκεί οι τροπολογίες. Το τελευταίο θέμα αφορά την πολιτική έβρεση τεχνιών. Και αυτό, κατά την άποψή μας, είναι πολύ σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω όμως ότι ακολουθούμε το σωστό δρόμο και ευχαριστώ θερμά τον κύριο Βίκνκλα για την μέχρι τώρα συνεργασία που είχαμε. Επόμενη παρεμβάση του κυρίου Τσουκαλά. Αλλά αν έχετε την καλοσύνη όλοι σας, μην ξεχνάτε το ρολόι η έκθεση του κυρίου Βίνκλερ παρουσιάζει αρκετές καλές προτάσεις για μια ευρεία ευρωπαϊκή στρατηγική για την καινοτομία που θα ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες ανάγκες. Με τις τροπολογίες που κατέθεσα θέλησα να προσθέσω και να τονίσω ορισμένα σημεία που θεωρώ ιδιαίτερο σημαντικά, όπως για παράδειγμα την ισότιμη θεώρηση και των τριών πτυχών του τριγώνου της γνώσης καθώς και τη στενότερη σχέση μεταξύ καινοτομίας και επιχειρηματικότητας μέσω της ενδυνάμωσης του διαλόγου πανεπιστημίων και επιχειρήσεων. Πρόσφατα ψηφίσαμε σχετική γνωμοδότηση της κυρίας Μαντουρέλ και τη στήριξη των πρωτοβουλειών δημιουργίας ειδικών ζωνών καινοτομίας και επιχειρηματικότητας γύρω από τα πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα. Σήμερα η Ευρώπη διαθέτει περισσότερες από 2.000 νησίδες, αλλά ελάχιστες από αυτές είναι παγκόσμιας εμβέλειας. Η αύξηση της παροχής κινήτρων είναι επίσης καθοριστική σημασίας για την προσέλευση όχι μόνο ερευνητών και ειδικευμένου προσωπικού εντός και εκτός Ευρώπης, αλλά και για την προσέλκυση επενδύσεων. Για το λόγο αυτό προτείνω με την τροπολογία μου 60 την ανάγκη διάθεσης του 10% της χρηματοδότησης κάθε ευρωπαϊκού προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Τέλος, πολύ σημαντικό σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που αναλαμβάνονται για την προώθηση της ευρωπαϊκής καινοτομίας είναι να υπάρχει μια περισσότερο ανθρωποκεντρική θεώρηση και κατά τη χάραξη στρατηγικής της καινοτομία, μιας και ο άνθρωπος αποτελεί την κινητήρια δύναμη όλων αυτών των προσπαθειών και από αυτόν εξαρτάται η επιτυχία των αποτελεσμάτων. Σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και έτσι αυτό το θέμα της σημερινής διάταξης ε, έκλεισε. Ο εισηγητής δεν θέλει να απαντήσει και νομίζω ότι στις 8 Απριλίου μπορούμε να ψηφίσουμε. Πάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι οι ψηφοφορίες. Ελπίζω να έχετε όλοι μαζί σας ε, τις ε, κάρτες σας για να ψηφίσετε. Ε, δεύτερον, να τις βάλετε μέσα στη σχισμή και αν συμφωνείτε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν με την έκθεση Τόγια.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 κατά αποχές εγκρίνεται ως εκ τούτου οι 46 έως το 48 καταπίπτουν πάμε 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε στην 55. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 57. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρούντε, ε, συγγνώμη, 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, με συγχωρείτε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Μισό λεπτό, την 59 να την ελέγξουμε. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 59. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εντάξει. Πολύ ωραία. Η 60. Υπέρ. Τι έγινε. Υπάρχει πρόβλημα. 19 κατά. Κυρία Μαντουρέλη.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 Λοιπόν, πρώτο τμήμα στην 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται.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 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 95 μισό λεπτό καταπίπτει λέει ο πρόεδρος. 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά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 αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος, ηλεκτρονικός έλεγχος για τη συμβαστική 4. Λοιπόν, 4α, συμβαστική 4α, για αυτήν ψηφίζουμε. τρεις του ΕΛΚ είναι παραπάνω από ό,τι προβλέπετε. Ε, μισό λεπτό. Έκλεισε η ψηφοφορία. Συν ένας, δύο, Μίστερ Μανουέλ, μισό λεπτό. Υπερψηφίζεται λοιπόν. Συμβαστική 4β καταπίπτει. Τσίτσεστερ. Ο Τσάρλς έχει το λόγο. Πρόεδρε, στην οθόνη βλέπουμε τον αριθμό όσων ψήφισαν και όσων υπερψήφισαν, αλλά όχι το σύνολο των πληροφοριών. Μήπως μπορείτε λιγάκι να βελτιώσετε τις πληροφορίες που αναγράφονται στον πίνακα. 29 συν 2, 31 συν και 20 ε, κατά. Εντάξει. Που σημαίνει ότι ε, η Β, η τροπολογία καταπίπτει, πάμε στην 116. Υπέρ 116 παρακαλώ. Κανείς. 116 ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 117 ε, ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 121 υπέρ κατά απορρίπτεται πάμε τώρα ε, στα ε, εκτιμώντας ένα υπαριθμόν ένα υπέρ για την 121 ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ ηλεκτρονικός έλεγχος για την 121, 121 ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε. 30 υπέρ, 19 ε, κατά. Εγκρίνεται. Λοιπόν, εκτιμώντας 1 υπέρ. Κατά. Πάμε τώρα ε, στα υπέρ για το 1, κατά, απορρίπτεται. 2, Κτιμώντα 2, υπέρ, όχι, όχι, ηλεκτρονικός έλεγχος για το 1, ηλεκτρονικός έλεγχος για το 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε. 27-20 εγκρίνεται. Τι έγινε με τους δύο που δεν έχουν ε, ε, κάρτα για να ψηφίσουν. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Πολύ ωραία. Εγκρίνεται. Για το δύο... τώρα ψηφίζουμε για το 2. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το 3 καταπίπτει για το 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, καλύτερα ε, ηλεκτρονικός έλεγχος. Παρακαλώ για το 5 άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Πάμε στο 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Οκτώ υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για το 8 άρχεται η ψηφοφορία έκλεισε μία ψήφος του ΕΛΚ ε, παραπάνω από ό,τι προβλέπετε,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 Πολύ ωραία λοιπόν, έκλεισε η ψηφοφορία. Αποτέλεσμα απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά, άποχες εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, άποχες απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 22 21 ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία Έκλεισε ναι, μισό λεπτό έκλεισε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 στην ε, γνωμοδότηση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Εκτιμώντας ένα της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Για άλλη μια φορά. Επανέλεγχος. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δύο. Καταπίπτει. Τρία του περιβάλλοντος, της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην 5, στην τελευταία μονοπρόταση, υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Στην 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Για το 5, μάλλον για το 10, ε, η τροπολογία 10, επανέλεγχος. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται η τροπολογία υπεριθμών 10. 15 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 20 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 21 καταπίπτει, 22 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 23 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 24 καταπίπτει. Πολύ ωραία λοιπόν. Ε, Ψηφίζουμε για το τελική ψηφορία ηλεκτρονική. Άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε. Πανέλεγχος. Πάλι ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Έκλεισε λοιπόν η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η έκθεση συγχαρητήρια. Επόμενο σημείο. Λένε Χεκ. κάποια ψηφορία πάλι. Πάω εδώ. Έκθεση ΕΚ. Σημείο 1. Ε, τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. ΕΝΒΙ NV11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρία συμβιβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Α, 37 και 38, συγγνώμη. 37 και 38 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ένβη 13. Α, όχι, 7. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. Είναι 13 τώρα. Υπέρ. Κατά. αποχέ, εγκρίνεται. 41. Με μια προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. NV16. NV16 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ Α, όχι, καταπίπτει το δεύτερο τμήμα, δεν έχει νόημα. Μάλιστα. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Κλοντ μα μήπως θα πρέπει να ψηφίσουμε την NV20 γιατί 56 δεν κρίθη. Ναι, ναι, ναι, ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι δεν είναι κρίθη 56. Λοιπόν, NV20 nv υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικός έλεγχος για την nv EPP too much. Δύο του ΕΛΚ περισσότερο από το πρέπει. Τώρα εντάξει, ωραία, πέρασε τι ψηφοφορίε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Και 15 ψηφίσαμε. NV22 υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Ενεκρίθη νομίζω, αλλά να ελέγξουμε. Έλεγχος από το 21. 21 λέω έλεγχος. Πέρας ψηφοφορίας. Ναι, ενεκρίθη πράγματι. NV2, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. NV3, υπέρ. Κατά. Αποχές. Είναι κρίθη. NV4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Είναι κρίθη. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Έλεγχος γιατί την 5. Άρχη ψηφοφορία. Πάλι δύο από το έλκυνο υπεράριθμοι. Πάντα ήδη φαίνεται. No? One EPP too much. Still. Okay. Ένας έτσι Α, ωραία τώρα. Εντάξει. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τριάντα τέσσερα. Τριάντα τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. οκτώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. NV8. Ελέγχουμε. Άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Μάλιστα. NV9. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Α, όχι. Δεν έχει νόημα. Να ελέγξουμε το πρώτο τμήμα της NV9. Να ελέγξουμε το πρώτο τμήμα της NV9. Άρχεται ψηφοφορία. Δεν εκριθη κρίθη. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. NV10. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Έλεγχος NV10. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Όχι, δύο έλκυνε υπεράριθμοι πάλι. Εντάξει τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Ενεκρίθη. 51 προς 1. Ωραία. Και περνάμε τώρα στο σημείο 8 της διάταξης. Ναι, συγχαρητήρια βέβαια. Ε, δεν χρειάζεται να το λέω κάθε φορά. Εγώ συγχαίρω όλους τους συζητητές, δύο εκείνους που έχουν θετικό αποτέλεσμα της έκθεσης. Περνάμε στην ε, ψηφοφορία 8, σημείο 8. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 39 καταπίπτει. 40 υπέρ. Κατά αποχές. Α, 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41 ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 καταπίπτει συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ 18 υπέρ λέω. Ξανά. 18 υπέρ κατά αποχές έλεγχος, ναι, έλεγχος. 18 ηλεκτρονικός έλεγχος, 18. Δύο και περάριθμε. Εντάξει, τώρα πέρασε η Είναι κρίθη. Δεκαεννέα, υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται 20 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 44 προσθήκη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48 Όσο προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 50 ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 51 πάλι έρθει προσθήκη. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 52 άλλη προσθήκη. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 καταπίπτει. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 28 πρώτο τμήμα έλεγχος. Άρχιψη φορεία. Ένας υπεράριθμος του ΕΛ. Εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28. υπέρ. Όχι, 58. ψηφίσαμε το 28.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 Πέρας πληροφορίας. Απερίφθη πράγματι. Πέμπτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30 σε δύο τμήμα. Πρώτο τμήμα. Πρώτο τμήμα 30 υπέρ. Κανένας. Ξανά. 30 πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Έλεγχος. Πρώτο τμήμα της 30. Άρχεται η ψηφοφορία. Ένας υπερόπτυμος του ΕΛΚ. Εντάξει τώρα, πέρας. Είναι κρίθη. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. εξήνθος προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 61. Υπέρ. Κατά. εποχές, Εγκρίνεται. Η κυρία Εκ. Για την 59 πρόεδρε. Λέει καταπίπτει αν εγκριθεί 30. Λένε ότι 30 δεν εγκριθεί όμως.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 αποχές απορρίπτεται. Υπάρχουν προβλήματα με τη διερμηνία, όχι ακόμα. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά χε συγκρίνεται, 2 υπέρ κατά χε συγκρίνεται, 35 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 καταπέψη 3 υπέρ υπέρ για την 3 κατά ξανά παρακαλώ τροπολογία 3 υπέρ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 Τελική ψηφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται. Two EPP too much, please. One too much. One PPT, one PPE too much. Ένας υπεράριθμος ακόμα του ΕΡ. Closed and it's adopted. 47 υπέρ, 5 κατά εγκρίνεται.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 αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 8 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ Α, 14, συγγνώμη. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Έλεγχος για 14. Άρχιε ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ένα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά έλεγχος για τη 2 έλεγχος για τη 2 πέρας φορές mm. εγκρίνεται 17 κατά δύο τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 18 ως προσθήκη υπέρ. Ορίστε. Δεν ακούτε πια. Some problems? We try it. Once again. με ακούς τώρα, εντάξει, ωραία. Ε, ναι, ευχαριστώ που με καταλαβαίνεις. μια ερώτηση για την προηγούμενη ψηφοφορία Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που ψηφίζουν χωρίς κάρτες ή όλοι ψηφίζουν με κάρτες. Γιατί έχω την εντύπωση ότι εάν κάποιοι ψήφιζαν χωρίς κάρτα, το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό. Πρόεδρος, να ευχαριστώ για την ένδειξη αυτή. Εγώ θεωρώ ότι εάν κάποιος δεν το πει, το αποτέλεσμα ισχύει οι συνάδελφοι που δεν έχουν κάρτα θα πρέπει για κάθε ψηφοφορία να μου το λένε. Δεν μπορώ εγώ να το ρωτάω, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι υπερβολικό. Εάν με Εάν κάποιο δεν έχει κάρτα, πρέπει να μου το πει. Και άλλο πρόβλημα. Θα ήθελα να ρωτήσω τη γραμματεία κατά πόσο υπάρχει επαρκής αριθμός σοσιαλιστών στην ψηφοφορία αυτή. Αν υπάρχουν αρκετοί σοσιαλιστές. Εμείς κοιτάμε τους υπεράριθμους. Τώρα αν λείπουν κάποιοι... Όταν δεν είναι ονομαστική ψηφοφορία, το μόνο που μπορούμε να ξέρουμε είναι αν υπάρχει κάποια ομάδα που έχει υπεράριθμους, αλλά όχι αν έχει λιγότερους. Gut, also das ist wichtig. Wir können hier... Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό. Ηλεκτρονικά βλέπουμε αν υπάρχουν υπεράριθμοι, όχι αν υπάρχουν ε, ελλειπείς, αν υπάρχει ελλειπής αριθμός. Και γι' αυτό έχει δίκιο ο Τσάρλς. Αν κάποιος θέλει να ψηφίσει χωρίς κάρτα, πρέπει κάθε φορά πριν από την ηλεκτρονική ψηφοφορία να το λέει. Δεν μπορώ να το σημειώνω εγώ κάθε φορά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η κυρία Μαντουέλ. Εγώ ψηφίζω χωρίς κάρτα, αλλά μου λένε ότι έχουμε επαρκή αριθμό, δηλαδή ότι εμείς έχουμε απαρτία αλλά θα ήθελα να με λάβετε υπόψη διότι δεν έχω την ηλεκτρονική μου ε, κάρτα. Τι Δηλαδή, θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτή την παρατήρηση του Τσάιλς. Εάν είναι στενή η πλειοψηφία, πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου. Αλλά τώρα πάει. Σημείο 3, εντάξει. Α, όχι το 18 πρώτα. Ναι, 18 πρώτα. Ποιος είναι υπέρ της 18. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος. Καλά. Να εγκρίνουμε. Είναι μια προσθήκη. Καλύτερα να το ελέγξουμε. 18. Ελέγχουμε τη 18. Δύο έκρη υπεράριθμοι. Να τους δώσετε εκεί κάποιους ψήφους στις ξέρω εγώ. Λοιπόν. τη πληροφορία. 20 προς 30. Και η κυρία Μαντουρέλ υπέρ ή κατά. Κατά. Ακόμη καλύτερα. Εντάξει. Δεν παίζει ρόλο. απερίπτει ούτως ή άλλως. Τρία, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται. Να μην έχουν πάρει αριθμούς ε, ΕΛΚ πάλι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Έκθεση Ζαϊκαρίν. Και δεν είναι η τελευταία ψηφοφορία αυτή τώρα. Έχουμε άλλη μια. Δεν προχωράμε πολύ γρήγορα σήμερα. Λοιπόν, ψηφίζουμε. 54, 54, 53, 63 και 203 on block. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 55 και 45. Υπέρ. Υπέρ λέω. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 56. Υπέρ. Έλεγχος. 55 και 45 on block ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Άρχιψη φορεία. Πέρας. 20 προς 28 κύριε Μοντουρέλ κατά. Α, απερίφθη. 56 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα, μπλοκ 58, 59, 60, 150, 151, 153, 154, 155, όλα μαζί. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 61, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται σε δύο τμήματα την 62. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Unblock 2, 3, 4 και 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Απεχές. Εγκρίνεται. 71. Υπέρ. Κατά. Απεχές. Εγκρίνεται. 72. Υπέρ. Κατά. Απεχές. Απερίπτεται. 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 76 και 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται 8 υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Εδώ. Αποχές. Εγκρίνεται. 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 82, 93 και 105. Υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 83. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 83. Closed. Rejected. Απορρίπτεται. 84. 84. Καταπίπτει. 84. Υπέρ. Κατά. 84. Ε, υπέρ, ε, ξανά παρακαλώ, το υπέρ για το 84. Κατά έλεγχος, ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Για το 84 έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 96 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 99 υπέρ, κατά, Έλεγχος ηλεκτρονικός. Για το 99 έκλεισε. Ε, απορρίπτεται. Το 100 και 101. Όλα μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ, κατά, αποχές, 108 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ε, ε, δεν είπε ο πρόεδρος αποχές, τέλος πάντων εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος ηλεκτρονικός. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το 15. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 112 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 119 και 142 και 89 και 88 ενσώματι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ. Το αποσύρατε. Όχι. 121. Για το 121 ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 128 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 καταπίπτει 130 ε, ψηφίζουμε μόνο για τη δεύτερη πρόταση πρέπει πρέπει να ψηφίσουμε για το σύνολο του 130 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 133 δεύτερη πρόταση υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 47 μισό λεπτό 47, 52, 139, 138 ενσώματι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στο 143 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ ηλεκτρονικός έλεγχος για το 27. Για το 27 ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία, έκλεισε. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 152 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 έχει καταπέσει 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 163 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται νομίζω το επόμενο είναι 174 υπέρ Ξέχασα το 167. Είναι εκτός μικροφώνου, κυρία. Δεν ακούμε τι λέει. Κοιτάξτε, υπάρχει μια σύγχυση στη διερμηνία. όταν καταπίπτει μία τροπολογία ε, δεν ε, το προλαβαίνουν οι διερμηνείς. Ε, πρέπει λοιπόν να το προσέξουμε αυτό. Γίνεται μια σύγχυση και νομίζω ότι αυτό ισχύει για όλους, δεν ισχύει μόνο για μένα. Η συντονίστρια των συσχολιστών μου είπε ακριβώς το ίδιο και νομίζω ε, θα ήταν καλό να προσέξουμε, να είμαστε προσεκτικοί, ε, να μην τρέχουμε πάρα πολύ όταν καταπίπτουν κάποιες τροπολογίες και προχωράμε ε, με άλμα. Πρόεδρος, εγώ προσπάθησα να είμαι λίγο πιο γρήγορος έχοντας κατά νου το ρολόι, την ώρα αν θέλετε ε, να σας λέω ακριβώς μεγαλύτερες λεπτομέρειες, αλλά θα χρειαστούμε περισσότερο χρόνο. Λοιπόν, καταπίπτουν τώρα όλες οι τροπολογίες μέχρι και την 166, εν μέρη διότι είναι ταυτόσιμες και εν μέρη διότι έχουν καταπέσει. Ε, πρέπει να ψηφίσουμε για την 167 γιατί είναι προσθήκη. Υπέρ παρακαλώ. Δεν έχετε διερμηνία εσείς. Μπράβο. Λοιπόν, ξανά. Πρόεδρος, ε, ίσως ε, λιγάκι πρώτο έτρεξα. Λοιπόν, 167 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 168 και 169 ε, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε από αυτόν. 170 ενίδη προσθήκης υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 172 και 173 καταπίπτουν. Πάμε στην 174. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 171 ως προστίκη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 175 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 176 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 177 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 178 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 180 υπέρ κατά αποχές Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 180 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε. Απορρίπτεται. Η 181 αποσύρθηκε, 182 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 183 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 184 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 185 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 186 Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο, η 186 είναι ταυτόσιμη και δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε από αυτή. 187 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 188 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 189 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 190 υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Καλύτερα ε, να έχουμε έναν ε, ηλεκτρονικό έλεγχο, άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 191 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ξανά. 191 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 192 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 193 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 194, δεν ψηφίζουμε ταυτόσημη, 195 παρακαλώ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 40 μισό λεπτό ηλεκτρονικός έλεγχος. 195 έλεγχος ηλεκτρονικός. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία και απορρίπτεται. Και πάμε στη 40. 40 λοιπόν. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 196 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 197 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται όχι. Μισό λεπτό. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Για την 197 παρακαλώ. Ως προσθήκη. Έκλεισε. Απορρίπτεται. Πολύ ωραία. 198 υπέρ. Κατά. Αποχές. Το ίδιο πρόβλημα πάλι. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Είναι πολύ πιο εύκολο. 198 άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 199 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 200 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, απορρίπτεται. 201 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 202 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 204 υπέρ. 204 ε, υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. 205 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 206 υπέρ. Κατά. Κατά παρακαλώ αποχές εγκρίνεται. 207 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 208 και 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1 εκτιμώντας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία Άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε. Και εγκρίθηκε η έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Τζαβέλα. Η κυρία Τζαβέλα θέλει να μιλήσει. Να πει δυο λόγια. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κυρία Τζαβέλα. Κύριε Πρόεδρε, Είχα μία πρόταση της τελευταίας στιγμής από τους σοσιαλιστές, συμβιβασμός 7, 4β. Έχει την ε, ίδια σημασία, αλλά έχει διατυπωθεί καλύτερα. Θέλετε να σας το διαβάσω. 4β, όπως προτείνουν οι σοσιαλιστές. Κοιτάξτε να το πούμε καλύτερα σε εκείνο το σημείο όταν θα έρθει το σημείο αυτό. Να το πούμε όταν θα έρθει το σημείο αυτό, όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, εντάξει. Και θυμίστε το να το ξεχάσω. Πάμε στην συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρία, υπέρ. Όχι, μισό λεπτό λέει ο πρόεδρος. Πρώτα η επτά, Πρώτα η επτά, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Είμαστε στο επτά, Στην τροπολογία επτά απορρίπτεται. Και μετά συμβιβαστική τρία λέει τώρα ο πρόεδρος. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. 12 υπέρ. Δεν θα τις διαβάζω τώρα όλες. 12 υπέρ. 12 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα καταπίπτουν πάλι 22, 25, 24 και πάμε στην συμβιβαστική 7 και τώρα κυρία Τζαβέλα έχει το λόγο. Παρακαλώ κυρία Τζαβέλα για την συμβαστική υπερθμών 7. το νέο κείμενο. Το νέο λοιπόν κείμενο έχει ως εξής υπενθυμίζει την σημασία των τρεχουσών διαπραγματεύσεων για τον τομέα ελευθέρου εμπορίου και ε, ενθαρρύνει τις χώρες UFM να εργαστούν για την εναρμόνιση των θέσεών τους στα πλαίσια του, των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ. Αν κατάλαβα καλά, η κυρία Τζαβέλα, η συγγήτρια, ε, προτείνει αυτό να είναι μια νέα συμβαστική πρόταση. Σωστό κυρία Τζαβέλα. Συμφωνούν όλες οι άλλες πολιτικές ε, ομάδες. Πολύ ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν για τη νέα συμβαστική πρόταση, την 7. Ποιο συμφωνεί παρακαλώ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κατόπιν τούτου πάμε στην συμβαστική 8. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πολύ ωραία Τώρα, έχουν καταπέσει μία σειρά τροπολογιών και πάμε στην τροπολογία υπαριθμών 21. Ε, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 26 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική ε, ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε. Εγκρίνεται λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Τζαβέλα, θερμά συγχαρητήρια και για το γεγονός ότι μπορέσατε τόσες πολλές τροπολογίες να τις ε, συνοψίσετε. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το υπαριθμόν 6. Όχι, όχι, λάθος, το τι έξι λέει ο πρόεδρος, το 12 πάμε. 2 επί κάνει 12, λέει χαριτολογώντας ο πρόεδρος. Πάμε στο 12, ε, πρόκειται για τον ε, παροπλισμό των ε, μονάδων πυρηνικού σταθμού. Η συγγήτρια είναι η κυρία Χάρμς, αν τώρα ε, κάνατε λίγη ησυχία, ίσως η συνάδελφος ε, κυρία Χάρμς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 Και τώρα έχει το λόγο μόνο η κυρία Χάρμς. Πολύ ωραία λοιπόν. Ε, σήμερα συζητάμε για τις ε, τροπολογίες της, ε, στην έκθεση σχετικά με τα κονδύλια για τον ε, παροπλισμό του Κόσλο Ντούι. Ε, σύμφωνα με την ενταξιακή συνθήκη πρέπει να παροπληστεί αυτός ο ποινικός σταθμός και τα κονδύλια πρέπει να διατεθούν εν μέρη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω λοιπόν ότι μετά από πάρα πολλές συζητήσεις που είχαμε εδώ στην Επιτροπή μας αλλά και συζητήσεις μεταξύ Σκιώδου Σιγητού και μου ε, δεν χρειάζεται, επειδή έγιναν όλα αυτά, δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειε τη έκθεση. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι το εξή. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η δική μου η πολιτική ομάδα πιστεύει ανεπιφύλακτα το γεγονός ότι είναι σωστό η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τον παροπλισμό των ε, ε, αντιδραστήρων 1, 2, 3 και 4 του Κοσλοντούι ε, πριν υπογραφεί η συνθήκη ένταξης. Σωστό λοιπόν το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε τη δέσμευση να συμμετάσχει ε, στο κόστος ε, για την απομάκρυνση των ε, αποβλήτων, των πυρηνικών καταλήπων. Νομίζω λοιπόν ότι μέχρι τώρα για το πρόγραμμα αυτό δεν δόθη ιδιαίτερα μεγάλος όγκος κονδυλίων. Θα ήθελα όμως να δράξω την ευκαιρία για να σας πω το πόσο ακριβώς συνέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να ε, επομιστεί και αυτή ένα μέρος του παροπλισμού. Ο, ε, τα κονδύλια, η οικονομική υποστήριξη προς τη Βουλγαρία από το 1999 μέχρι το 2003 αυξήθηκε σημαντικά. Μιλάμε για 155 εκατομμύρια ευρώ από το 2004 μέχρι το 2006, 185 εκατομμύρια ευρώ και από το 2007 μέχρι το 2009 διατέθησαν 200 ε, τόσα εκατομμύρια ευρώ που σημαίνει συνολικά μέχρι την ε, επόμενη παρτίδα που θα, για την οποία θα πρέπει να αποφασίσουμε εκταμιεύθηκαν 550 εκατομμύρια ευρώ από τον κοινοτικό κορβανά προς τη Βουλγαρία. Και θέλω λοιπόν να διευκρινίσω το εξής. Επειδή αυτό προκάλεσε πάρα πολλές συζητήσεις στους σκιώδεις συγητές, ε, κυρίως, ο συνάδελφος κύριος Ρανστόρφ δεν ήθελε να με πιστέψει, αυτά τα χρήματα, τα 550 εκατομμύρια ευρώ, τα χρήματα αυτά εκταμιεύθηκαν σύμφωνα με την συνθήκη ένταξης της Βουλγαρίας. Έτσι λοιπόν αυτό το ποσό για το οποίο θα ψηφίσουμε αργότερα και στην Ολομέλεια, το ποσό αυτό αποτελεί ε, μια επιπρόσθετη οικονομική ε, χρηματοδότηση η οποία όμως δεν προβλέπεται στην αρχική, στις δεσμεύσεις μας. Από το 2010 μέχρι το 2013 θα διατεθούν κάποια κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη Βουλγαρία. Μιλάμε για 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το πρότεινε η Κομισιόν και εγώ ως εισηγήτρια ευθύ εξ αρχής ε, είπα ότι κατά την άποψή μας το, ποσοστό, το ποσό αυτό είναι ικανοποιητικό. Ε, σύμφωνα με την άποψη Κομισιόν τα 180 εκατομμύρια θα διατεθούν για τις ε, δραστηριότητες παροπλισμού αλλά και για την διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων γιατί είναι απολύτως απαραίτητο ε, να επενδυθούν χρήματα σε ενδιάμευσους ε, αποθηκευτικούς ε, χώρους για τα πυρηνικά κατάλοιπα. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει ακόμα στη Βουλγαρία. Εγώ λοιπόν Θεωρώ ότι για την διαχείριση των αποβλήτων και την τελική απομάκρυνσή τους, ε, επειδή ασχολήθηκα με το θέμα αυτό, καταλήγω στο ότι πραγματικά εδώ ε, πρόκειται για μια ανομαλία. Ναι μεν η Βουλγαρία ε, τάσεται ανεπιφύλακτα υπέρ της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας, το έκανε και εξακολουθεί να το κάνει και αυτή τη στιγμή αυτό, όμως μέχρι τώρα δεν έχει λάβει κανένα απολύτως μέτρο έτσι ώστε να μεριμνήσει για την τελική απομάκρυνση των ραδινεργών καταλήπων. Δεν υπάρχει καμία πολιτική για την απομάκρυνσή τους. Και ως εκ τούτου και ο Σκιώδης εισηγητής και εγώ καταλήξαμε στο ότι υπάρχουν ε, συμβάσεις με τη Ρωσία η οποία Ρωσία ε, θα δεχθεί, μας είπανε, ε, τα κατάλοιπα, τα ποινικά κατάλοιπα από τη Βουλγαρία. Το έκανε αυτό στο παρελθόν και ποτέ θα συνεχίσει να το κάνει και δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Αυτό μας είπαν. Και εγώ χαίρομαι για το ότι ο Επίτροπος Ενέργειας, ο κύριος Ότεγκερ, πήγε στη Βουλγαρία και κατόπιν τούτου επιτόπου στη Βουλγαρία κατέστησε σαφές ότι η εξαγωγή ιδιαίτερα υψηλών ραδινεργών καταλήπων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό δεν είναι αποδεκτός ε, τρόπος. Επίσης χαίρομαι για το ότι ο κύριος Ότιγκερ τους τελευταίους μήνες ανέφερε επανειλημμένα ότι ένα από τα βασικότερα προγράμματα με τα οποία ασχολείται ε, έχει ως στόχο να κατατεθεί μια οδηγία η οποία θα μεριμνεί για την ε, προετοιμασία και για την ε, δημιουργία ε, αποθηκών για πυρηνικά κατάλοιπα. Και αυτό αφορά κυρίως τα υψηλά ραδιενεργά κατάλοιπα. Η όλη διαδικασία, όπως σας είπα, έχει δρομολογηθεί και με, ε, εγώ περιμένω με μεγάλη υπομονησία αυτή την οδηγία. Δυστυχώς, Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το τέταρτο τμήμα των χρημάτων που προωθούνται προ την Βουλγαρία. Κατά τη γνώμη μου θα ήταν καλό να μπορούσαμε να είχαμε μπορέσει να το κάνουμε γιατί επιμένω ότι πραγματικά έχει φτάσει πια η ώρα στην Ρουμανία να μην εξά... στη Βουλγαρία συγγνώμη, να μην εξάγονται μόνο ε, τα απόβλητα αλλά να προετοιμαστεί η τελική αναπόθεση των αποβλήτων. η μόνη διαφορά που έχω εγώ είναι για την χρήση των χρημάτων που προωθούνται προς την Βουλγαρία. Θεωρώ ότι το επόμενο αυτό ποσό των 300 εκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2010-2013 εν μέρη θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν άμεσα για το Κοσλοντούι. Αυτό που προβλέπτω στα 180 εκατομμύρια των παραπλησμό, που φαίνεται ότι είναι ένα καλό ποσό και θα πρέπει ιδίω να χρησιμοποιηθεί για την υποδομή της προσωρινής συναποθήκευσης. Τα υπόλοιπα χρήματα, τα 120 εκατομμύρια δηλαδή, και αυτό είναι το κεντρικό σημείο της έκθεσής μου, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένες εργασίες για την προετοιμασία της τελικής ε, εναπόθεσης. η Βουλγαρία θα πρέπει να προσανατολιστεί σε καλές ε, πρακτικέ σε ευρωπαϊκές κοινωνικέ χώρες και επιγειτονικέ, όπω παραδείγματο είναι η Ελβετία και η Σουηδία που έχουν καλά πρότυπα για την τελική αποθήκευση. Δεν υπάρχει λόγος να φοβούμαστε ότι τα 127 εκατομμύρια δεν θα υπάρχει δυνατότητα να δαπανηθούν για την τελική αποθήκευση. Το θέμα είναι πότε θα αρχίσει πραγματικά η Βουλγαρία να αντιμετωπίσει αυτό το σημαντικό πρόβλημα της τελικής αποθήκευσης. Σε αυτό το σημείο και πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτηση και οδηγηθούμε προσεχώς στην ψηφοφορία για την έκθεση αυτή, θα ήθελα να έχω μία γνωμοδότηση από την Κομισιόν, μία αξιολόγηση της πραγματικής κατάστασης προετοιμασίας των, τελικών, των χώρων συγγνώμη, τελικής αποθήκευσης στη Βουλγαρία και θα χαιρόμουν εάν οι εκπρόσωποι της ε, Κομισιόν μπορούσαν να αναφερθούν στο ερώτημα που τίθεται συνεχών κατά πόσο τα 300 εκατομμύρια αυτά ευρώ είναι μέσα στα πλαίσια της ε, συνθήκης ένταξης, είναι εκτός, γιατί ε, ο συνάδελφος Ράνστορφ έχει μια τελείως διαφορετική άποψη που την έχει προωθήσει πολύ έντονα και έχουμε και δύο περαιτέρω βασικά θέματα που συζητήθηκαν ε, μεταξύ των εισηγητών και εδώ και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος χωρίς να μπορέσει να βρεθεί η τελική λύση. Κατά πόσον υπάρχει έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας στην Βουλγαρία. <clears throat> Γιατί μετά τον παραπλησμό των μπλοκ 2 και ένα και δύο, οι εξαγωγές ε, ηλεκτρικής ενέργειας από τη Βουλγαρία αυξήθηκαν τόσο σημαντικά και πώς μπορείτε να ερμηνεύσετε τις αυξανόμενες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά πόσον σχετίζονται άμεσα με τον παρεπλισμό του Κοσλοντούι. Αυτά εισαγωγικά. Νομίζω ότι μεταξύ των σκιωδών εισηγητών εξετάσαμε τα άλλα θέματα και είδαμε κατά πόσο είναι δυνατόν ή αδύνατο να υπάρχουν συμβιβαστικές λύσεις. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριο Ζήμπη και η κυρία Χέρτσοκ έχουν ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την Κομισιόν, η οποία συνεπώς κινείται προς μια κατεύθυνση που υποστηρίζει και το Κοινοβούλιο, δηλαδή όσον αφορά την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του τομέα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δημιούργησε τη βάση γι' αυτό το έτος 2002, ότι η προστασία από επικίνδυνες ε, ακτινοβολίες είναι αρμοδιότητα του Ευρωπαίου νομοθέτη όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια. Και η οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια του έτους 2009 αποτελεί εν τελευταία λύση τη βάση ε, για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου που αποκτήσαμε. Εκεί προβλέπεται η έγκριση βέβαια των ε, σταθμών πυρηνικής ενέργειας, αλλά συμπεριλάβατε και το θέμα του παρεπλισμού και τη νομική βάση για την αντιμετώπιση των αποβλήτων. Και η συνθήκη της Λισαβόνας μας δίνει στον τομέα αυτό αρμοδιότητες, ούτως ώστε να αποφεύγεται στρέβλωση των οργανισμού στον τομέα αυτό μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχουν ενιαία πρότυπα δηλαδή που είναι μια σημαντική πρόοδος κατά τη γνώμη μου και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν, ιδίω τον Επίτροπο Έτινγκερ, ο οποίος προανήγγειλε ότι κατά τον παραπλισμό και αποξήλωση ε, των πυρηνικών σταθμών και την τελική αποθήκευση των αποβλήτων να υπάρχουν ενιαία πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, στον uh, Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα είμαι ιδιαίτερα σύντομη. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο ζητήματα. Το ένα είναι ότι υπάρχει έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία δεν, είναι, δεν μας απασχολεί το θέμα κάθε αυτό, αλλά στα Δυτικά Βαλκάνια υπάρχει έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας που δημιουργεί πρόβλημα όχι μόνο για τη Βουλγαρία αλλά και για τις γείτονες χώρες. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρική ε, ενέργεια χωρίς προσυμφωνία. Άρα υπάρχει πρόβλημα αφότου έκλεισε το Κοσλοντούι και ιδιαίτερα για τα Δυτικά Βαλκάνια και χώρες απομακρυσμένες σχετικά. Όλες οι γείτονε χώρες έχουν, αντιμετωπίζουν μείζον πρόβλημα λοιπόν. Τώρα, ως προς το περιεχόμενο, το 2006 η Βουλγαρία δεν ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν η πολιετής χρηματοδοτική συμφωνία αποφασίστηκε. Γι' αυτό η Βουλγαρία δεν μπορούσε να ήταν μέλος και τότε η Επιτροπή Ήτρε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκριναν ότι παρόλα αυτά θα πρέπει να δοθεί παρόμοια βοήθεια στη Βουλγαρία ε, σε σχέση με τη Λιθουανία και τη Σλοβακία. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή πρωτοβουλία διότι οι τρεις χώρες αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε ομοιόμορφη βάση. Το 2006 όταν αποφασίστηκε η σε χρηματοδοτική βοήθεια ε, δεν ήταν μέλος η Βουλγαρία και γι' αυτό αντιμετωπίζουμε μείζον πρόβλημα από πλευράς ε, προϋπολογισμού. Άρα η Επιτροπή Ήτρε θα πρέπει να είναι ενωμένη επί του θέματος. Γιατί το αναφέρω αυτό γιατί φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία. Αυτό αληθεύει, αλλά εγώ ως εισηγήτρια για τον προϋπολογισμό του 2011 είχα ε, αποστείλει μια επιστολή στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και ένα από τα βασικά σημεία ήταν αυτή η έκθεση, ζητώντας δηλαδή τα χρηματοδοτικά μέσα. Και αυτό το αναφέρω διότι ο Σκιώδης του Υπροπολισμού 2011 από τους Πράσινους έχει μία εντελώς διαφορετική γνώμη ε, σε σχέση με, την, ε, με αυτή της κυρίας Ρεμπέκα Χάρμς. Θα ήθελα λοιπόν να είμαστε ενωμένοι και συνεκτικοί ζητάμε χρήματα. Θα πρέπει να είμαστε συνεπείς και σε παρόμοιες εκθέσεις. Θα ήθελα να το αναφέρω αυτό διότι δεν θα είναι τόσο εύκολο να κρατήσουμε αυτή τη θέση μέσω Επιτροπής Προϋπολογισμών. Όχι εξαιτίας του Κοσλοντούι, αλλά των μεγάλων προκλήσεων ως προς την ενδιάμεση αναθεώρηση της πολιετούς χρηματοδοτικής συμφωνίας. Θα ήθελα λοιπόν όταν μιλάμε για αυτή την έκθεση όλοι να συμβαδίζουμε και στη, στο προσχέδιο προϋπολογισμού, γιατί είναι ζωτική σημασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο σκιώδης ηγητής ο Σόρας έχει το λόγο. Köszönöm, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy eh, nagyon Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σημειωθεί το εξής. Έχω αρκετή κατανόηση για την ε, Βουλγαρία και μου φαίνεται ότι είναι σημαντικό να ενισχύσουμε αυτά τα σχέδια παροπλισμού. Στη Σλοβακία, στους αρχιπούχονες, έχουμε αρκετές εμπειρίες λέξη. Υπήρχαν πολλά προβλήματα και εκεί και γι' αυτό πιστεύω ότι στο μέλλον θα πρέπει να είμαστε πιο ισορροπημένοι στην αντιμετώπιση του θέματος παροπλισμού σταθμών πυρηνικής ενέργειας. Επειδή έχουμε υψηλά κονδύλια και τα χρήματα αυτά θα ήταν ίσως καλό να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση της ασφάλειας. Γιατί και ο παραπλησμός μέχρι στιγμής κόστησε αρκετά χρήματα και βλέπουμε ότι τώρα θέλουμε να επενδύσουμε ακόμα περισσότερα. Και θεωρώ ότι υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα γιατί ένα τμήμα των χρημάτων αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα φτάσουν στη Βουλγαρία, αλλά θα φτάσουν στη Ρωσία. Η Ρωσία είναι εκείνη που θα ωφεληθεί από τα χρήματα αυτά και θα πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη, γιατί είναι πολύ, πολύ απίστευτο θα έλεγα πόσα χρήματα κοστίζει ο παραπλησμός και πού προθούν τα χρήματα αυτά. Θα ήταν καλύτερα λοιπόν να υποστηρίξουμε την επίλυση του προβλήματος του τελικής αποθήκευσης στις χώρες μας για να έτσι να φροντίσουμε καλύτερα για την τροφοδότηση με ενέργεια. Πρώτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώνει εδώ ο κατάλογος ε, εμβάσεων, γιατί έχουμε και άλλα δύο θέματα που πρέπει να εξετάσουμε. Ο Στένος για ο σχεδοσυχητής έχει το λόγο. господин Ευχαριστώ. Σήμερα μας ε, απασχολεί αυτή η έκθεση και οι τροπολογία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που είχαν μια πολύ επικοδομητική προσέγγιση και που επιβεβαιώνουν την ανάγκη επιπρόσθετης ε, χρηματοδοτικής στήριξης για τον ε, παροπλισμό των ε, αντιδραστήρων που έχουν απομείνει και που υποστηρίζουν τον πυρηνικό τομέα στη Βουλγαρία. Θα πρέπει να αυξήσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς και τη χρήση πηγών, ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τον επιπρόσθετο εξυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα. Ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε παροπλήσει τέσσερις ε, αντιδραστήρες, τέσσερις δηλαδή πυρηνικές μονάδες μέχρι τώρα κάτι το οποίο σημαίνει πολύ ε, μεγάλες απώλειες από ενεργειακής πλευράς. Και μέχρι το 2009 και εξαιτία της βοηθείας Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάσαμε σε μία απόδοση της τάξης του ενός τρίτου. Άρα θα πρέπει να συνεχίσει η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε φορά που παροπλίζονται αντιδραστήρες ε, δεν αντιμετωπίζουμε ενεργειακή κρίση στη Βουλγαρία και αυτό οφείλεται στην αρρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο θα πρέπει να τονιστεί. Έτσι, μπορούμε να αποτρέψουμε μελλοντικές ε, κρίσεις. Εάν αντιμετωπίζαμε μια τέτοια ενεργειακή κρίση, θα έπρεπε να ανοίξουμε εκ νέου τους αντιδραστήρες. Και αυτό είναι μια ρήτρα η οποία εγγράφεται στη συνθήκη προσχώρησης της ε, Βουλγαρίας. Ένα βασικό πρόβλημα στην πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγκυται στη θέση των πρασίνων, διότι θεωρούν ότι το 40% της επιπρόσθετης χρηματικής βοήθειας θα πρέπει να ε, στραφεί στην αναβάθμιση του συστήματος και στην προσωρινή, στις προσωρινές αποθηκεύσεις. Ε, δεν εγκρίνουμε κάτι τέτοιο, διότι τώρα η Βουλγαρία έχει μία διαφορετική στρατηγική για τη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων Πρόκειται για μια επιχειρησιακή στρατηγική που είναι, πολύ, που είναι γνωστή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ευρέως γνωστή σε όλες τις χώρες για την ε, διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων. Σύμφωνα με αυτή τη στρατηγική, εμείς προτιθέμεθα να ε, να αποβάλουμε και να αποθηκεύσουμε τα ε, ακτινοβολημένα αυτά απόβλητα. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί από τη μία μέρα ε, στην άλλη. Θα συμβεί κατά τα επόμενα χρόνια, αλλά βαθμία. Και με βάση την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασχολούμαστε ασχολούμαστε με την προσωρινή αποθήκευση πυρηνικών αποβλήτων, δημιουργούμε τέτοιες μονάδες για τα επόμενα 100 χρόνια. Αυτή είναι η προσέγγιση, αυτή η προσέγγιση μας και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την, ε, τις ανάγκες των εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η χρηματική βοήθεια θα χρησιμοποιηθεί για να ε, χτίσουμε αποθηκευτικούς χώρους για, να, για τα πυρηνικά απόβλητα. Τώρα, ένα 40% όπως ήταν η πράσινη να το ε, στρέψουμε προς μία άλλη κατεύθυνση δεν μπορεί να γίνει. Είναι κάτι το οποίο δεν σχετίζεται με τον παροπλισμό των τεσσάρων μονάδων. Για να γίνει κάτι τέτοιο, αν γίνει κάτι τέτοιο, πιστεύω ότι θα οδηγήσει στο μπλοκάρισμα αυτών των χρημάτων για μακρά χρονικά, χρονική περίοδο, κάτι το οποίο είναι αντιπαραγωγικό και δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε. Dovolte mi, ευχαριστώ, Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια όταν ορίζει ψηλά πρότυπα στην αποθήκευση των πυρηνικών αποβλήτων και στις προσπάθειές της για την ε, ασφάλεια. Από μεριά, πώς το βλέπουμε το θέμα της ε, οριστικής αποθήκευσης στην ε, ρωσική επικράτεια. Εμένα δεν με σοκάρει το γεγονός ότι πρόκειται να γίνει εκεί, γιατί εμάς που αυτό που σε ενδιαφέρει είναι να γίνει ασφαλής η αποθήκευση, άσχετα που θα γίνει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την κατάσταση μιας νέας ε, χώρας μέλος που έχει να αντιμετωπίζει αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα. Η τσεχική ε, δημοκρατία ήταν η μόνη που κατάφερε να διατηρήσει τις επενδυτικές της μονάδες στην ίδια κατάσταση όπως εκείνη που ήταν πριν από την ένταξη. Οι, οι Σλοβάκοι φίλοι μας δεν είχαν δυστυχώς την ίδια επιτυχία. Ε, έχω να πω ότι κυρίως τα προβλήματα ήταν πολιτικής μορφής, όχι τεχνολογικής και γι' αυτό μου φαίνεται περίεργο όταν εξετάζουμε ότι παραδείγματο χάρη η Βουλγαρία εξάγει περισσότερο, περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από πηγές οι οποίες όμως οδηγούν σε υψηλότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δεχθούμε και το γεγονός ότι στα δυτικά Βαλκάνια υπάρχει έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας σημαίνει ότι ακριβώς είναι οι επιπτώσεις αυτές από την παραπλησμό του Κοσλοντούι. Πρόεδρε, θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω για τις προσπάθειες που ε, αναλαμβάνονται. Θα ήθελα να αναφερθώ στις τρεις χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα. Δεν τη ζηλεύουμε καθόλου, διότι από το 2001 τα πολιτικά κόμματα αλλά και ο μέσος άνθρωπος ε, θα πρέπει να, μάλλον τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να επεξηγήσουν αυτό το θέμα στον απλό πολίτη. Είναι δυσνόητο βεβαίως και στη Λιθουανία αντιμετωπίζουμε αύξηση των ενεργειακών τιμών κατά 15%. Νομίζω ότι το ίδιο σενάριο ισχύει και για τις άλλες δύο χώρες. Υποστηρίζω ορισμένες τροπολογίες, ιδιαίτερα εκείνες που τονίζουν το ρόλο του EBRD και την χρηματοδότηση του παροπλισμού. Νομίζω ότι το ελεγκτικό συνέδριο θα πρέπει να ελέγξει ορισμένα στοιχεία εδώ και ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που έθιξε ο εισηγητής είναι η διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων. Νομίζω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προβάλλει μια πρόταση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα στο μέλλον, διότι είναι ένα λεπτό κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Η Λιθουανία αυτή τη στιγμή ε, κατασκευάζει αποθηκευτικούς χώρους και μονάδες. Το ίδιο κάνει και η Βουλγαρία, αλλά αυτό δεν αρκεί για το μέλλον. Γι' αυτό θα πρέπει να αρχίσουμε να το συζητάμε τώρα. Υποστηρίζω το συνάδελφο που λέει ότι θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι διότι είναι ένα πολύ ε, ευαίσθητο πολιτικά ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξαναδώσω το λόγο στην ισχύτηρη κυρία Χάμς. Παρακαλώ να είναι πάρα πολύ σύντομη, γιατί πραγματικά δεν έχουμε χρόνο. Ναι. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι λυπάμαι που ο εκπρόσωπος της Κομισιόν δεν πήρα το λόγο. Α, όχι, θα τους δώσω το λόγο, θα τους δώσω το λόγο. Είχατε ζητήσει το λόγο εσείς. Α, Θα προτιμούσα να μιλήσω στο τέλος, Πρόεδρε, ίσως να ακούσουμε πρώτα την Κομισιόν. Α, εγώ ήρθα σε κάτι που είχα ζητήσει το λόγο και δεν ήθελα να μη σα τον δώσω. Παρακαλώ, ο Διευθυντής κ. Φάρος έχει το λόγο. Ε, <clears throat> ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βέβαια θα αναφερθούμε στα άμεσα ερωτήματα και στην εξήγηση της πρότασής μας. Το σημείο εκκίνηση όσον αφορά τη χρηματοδότηση είναι καταρχήν το εξή. Μετά, μέσα στα πλαίσια τη ε, συνθήκη ένταξη της Βουλγαρίας είχε εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση μέχρι το 2009. Από την άλλη μεριά, για τη Λιθουανία και τη Σλοβακία η χρηματοδότηση είχε εξασφαλιστεί μέχρι το έτος 2013. Σημαίνει αυτό ότι αν θέλουμε να θέσουμε επίσης όρους τους Βουλγάρους, ε, τους ε, ε, Λιθουανούς και τους Σλοβάκους, χρειαζόμαστε μια νέα πρόταση για να καλύψουμε τα έτη 2010-2013. Αυτή είναι ακριβώς η πρόταση που έχετε μπροστά σας. Το δεύτερο σημείο είναι το σημείο της διαφοράς μας με την εισηγήτρια, που θα είμαι σύντομος. Εδώ εξετάζεται το θέμα, τα χρήματα του δεύτερου τμήματος, τα 120 εκατομμύρια πώς θα χρησιμοποιηθούν για ενεργειακά μέτρα ή για μέτρα για ένα τόπο τελικής αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων. Λυπούμε που ε, υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πρόταση για την τελική αποθηκευσή η οποία δυστυχώς χρειάστηκε να γίνει γιατί ήμασταν υπό πίεση χρόνου αλλά βάσει των εργασιών της Κομισιόν που υπάρχουν και στη διάθεση του Κοινοβουλίου και μετά τις προαναγγελίες του Προέδρου Παρόζο και του Επιτρόπου Έντιγκερ, είναι σαφές ότι η Κομισιόν σκοπεύει στο δεύτερο ημισή τρέχοντος έτους να υποβάλει μία πρόταση για την τελική αποθήκευση των ε, πυρηνικών αποβλήτων. Η πρόταση αυτή θα αναφέρεται βέβαια και στο θέμα της τελικής, τελικής αποθήκευσης. Μέσα στα πλαίσια του Κοσλοντούι αν εκεί ληφθεί μία απόφαση για τα απόβλητα θα προδικάσει βέβαια τη δική μας πρόταση. Ε, θα υπάρχει ζήτηση για τη χρηματοδότηση τελικών ε, χώρων αποθήκευσης και θα τίθεται το θέμα γιατί μέσα στα πλαίσια ε, του θέματος αυτού τελικής αποθήκευσης δίνουμε προτεραιότητα στη Βουλγαρία. Εμείς ε, θεωρούμε ότι θα ήταν καλύτερα να χρηματοδοτήσουμε τα 120 εκατομμύρια ευρώ αυτά σε μέτρα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι δύο μονάδες που έχουν παραπληστεί ξεπερνάνε το δυναμικό που θα χρειαζόταν. Εκτός αφήσεις, το... οι δυνατότητες παραγωγής στη Βουλγαρία διαφέρουν πάρα πολύ και μέσα στα πλαίσια των δικτύων διανομής υπάρχουν ανάγκες επένδυσης. Όλοι ξέρουν πια πόσο μεγάλη ζήτηση ενέργειας έχει η Βουλγαρία που ξεπερνάει τον κοινοτικό μέσο όρο. Έτσι χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα αποτελεσματικής χρήσης της ε, ε, ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα αυτή. Και αυτό διαφαίνεται και στην έκθεση της εισηγήτριας. Η κατάσταση στην ε, Βουλγαρία είναι ότι δεν υπάρχει έλλειψη τώρα, αλλά ότι μειώθηκαν οι εξαγωγές ε, στην περιοχή. Εκτός αυτού, η αντικατάσταση της παραγωγής των τεσσάρων αντιδραστήρων γίνεται από συντηρητικές ε, μονάδες σε μεγάλο ποσοστό οι οποίες βέβαια παράγουν διοξείδιο του άνθρακα και γι' αυτό έχει υπάρξει τεράστια αύξηση των εκπομπών διοξείδιου του άνθρακα. Η αναφορά στο ηλεκτρικό συνέδριο. Εμείς υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία του ηλεκτρικού συνεδρίου που αυτή τη στιγμή ακριβώς οργανώνει μια ακρόση των προγραμμάτων και για τα τρία κράτη, Λιθουανία δηλαδή, Σλοβακία και Βουλγαρία. και ως ε, Κομισιόν είχαμε ζητήσει και έλεγχο ε, της χρηματοδότησης ε, για το πρόγραμμα Μπούλιτσε και η επόμενη συνεδρίαση των χρηματοδοτούντων θα ενημερωθεί για τα αποτελέσματα αυτής, αυτού του ελέγχου του δημοσιονομικού και λογισμικού ελέγχου. Κατά τα άλλα, ευχαριστούμε την κυρία Χάρμς για την υποστήριξή της. Θεωρούμε ότι τα 120 εκατομμύρια για μέτρα παραγωγής ενέργειας ή αποτελεσματικής χρήσης ενέργειας είναι λογικά, γιατί πιστεύουμε ότι αυτού του τύπου τα προγράμματα θα πρέπει κατά τον ίδιο τρόπο να χρηματοδοτηθούν με το 2013 στη Λιθουανία και στη Σλοβακία. Αν θέλουμε λοιπόν να αναφερθούμε σε ίση μεταχείριση των τριών χωρών, υπάρχει νόημα και στη Βουλγαρία μέχρι το 2013 να ενισχύσουμε μέτρα ενεργείας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ η κυρία Χάρμς έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ την ε, παρουσίαση του εκπροσώπου της Κομισιόν. Ήταν πάρα πολύ καλή η συνεργασία με την Κομισιόν και όσον αφορά την προετοιμασία της έκθεσης και τα αριθμικά στοιχεία που είχαμε στη συζήτηση στοιχεία τα οποία προέρχονται από τις ανακοινώσεις κομισιών. Θα ήθελα εγώ να αναφερθώ σε δύο θέματα που με απασχολούν και τώρα και πέρα από τη ψηφοφορία. Εν μέρη με σοκάρει το γεγονός πόσο φυσιολογικό θεωρείται να μεταφέρονται τα απόβλητα αυτά για επανεπεξεργασία και τελική αποθήκευση στην Ρωσία, χωρίς να εξετάζεται πόσο επιβαρύνεται η υγεία των ε, κατοίκων εκεί και το περιβάλλον. Και ευχαριστώ όλους αυτούς που είπαν πραγματικά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στην διάγουσα και ε, κάνω έκκληση ιδίως στους συναδέλφους από τη Βουλγαρία να ασχοληθούν πολύ περισσότερο και πολύ πιο έντονα με το θέμα αυτό, ούτω ώστε ήδη σήμερα η ευθύνη για τα πυρηνικά απόβλητα που παράγονται στην ίδια χώρα και είπατε, πολλοί κέρδισαν αρκετά χρήματα με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και συνδυατή τη Βουλγαρία. Θα πρέπει έγκαιρα να γίνουν δεκτά αυτά τα στοιχεία που αναφέρονται γιατί κανένας δεν είχε αναφερθεί μέχρι στιγμή πώς θα γίνει η τελική αναπόθεση ιδίω του πυρηνικού, των πυρηνικών στοιχείων που βρίσκονται ακόμα σε ενεργή ακτινοβολία. και έτσι και στο Κοσλοντούι και στην Μπουγνίστα και στην Ζιναλίνα υπάρχει ακριβώς ο στόχος με τα χρήματα αυτά να εγγυηθούμε την ασφάλεια των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα απόβλητα τα αποστέλουμε στη Ρωσία. Και καταρχήν με απασχολεί και το θέμα γιατί στις νέες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τόσο έντονη έντονος ο φόβος της εξάρτησης από τις εισαγωγές φυσικού αερίου από την Gazprom. Από την άλλη μεριά δεν υπάρχει κανένας φόβος ότι ίσως στον τομέα της πυρηνικής υποδομής θα είμαστε απόλυτα εξαρτημένοι από την Ρωσία. Γιατί ο ε, πουλάει πολύ υλικό. Όχι μόνο στη Βουλγαρία, η Ρουζατρόμ εξετάζεται και σαν ε, παραγωγός νέων μονάδων, κατασκευαστής νέων μονάδων. Έτσι μπορούμε να αποφύγουμε στα νέα κράτη-μέλη την εξάρτηση, έτσι μπορούμε να έχουμε τη μεγαλύτερη α, εξάρτηση, γιατί όπως το ξέρω η Ροζατόμ είναι 100% θηγατρική της Κάσπρο Και κατά τη γνώμη μου, αυτό που γίνεται είναι ότι συνεχίζονται κάποιες παλιές εξαρτήσεις και δεν οδηγούμεθα σε ανεξαρτησία αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα μπορέσουμε να συζητήσουμε περισσότερο όταν ο κύριος Έτυγεν υποβάλει την πρόταση οδηγία. Και δεν μπορώ παρά να ελπίσω ότι θα είναι τόσο φιλόδοξη η πρόταση αυτή όσο υποσχέθηκε ο κύριος Έτυγεν ότι η ασφάλεια θα είναι το πρώτο, η ασφάλεια θα είναι το δεύτερο, η ασφάλεια θα είναι το τρίτο σημαντικό στοιχείο που θα ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και προσβλέπω με ενδιαφέρον στην ψηφοφορία. Πάμε λοιπόν ε, στο επόμενο θέμα. Έχουμε άλλα δύο θέματα, δύο εισηγήσει. Η κυρία Φιγκερέρα είναι εισηγήτρια και θα ήθελα παρακαλώ να δώσω το λόγο. Με την παράκληση, αν έχει την καλοσύνη, να χρησιμοποιήσετε μόνο 10 λεπτά και ο επόμενο εισηγητή και αυτό άλλα 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Η έκθεση αυτή που καταρτίζουμε στα πλαίσια της Επιτροπής Απασχόλησης μας οδήγησε σε μία ε, γνωμοδότηση η οποία θα πρέπει να καταρτιστεί σύμφωνα με όσα προτείνει η Ήτρε γενικότερα για αυτά τα ζητήματα. Σήμερα ήδη έγιναν ορισμένες συζητήσεις για να φτάσουμε στην απότερη κατάρτιση αυτής της γνωμοδότης. Χωρίς μικρόφωνο η ομιλήτρη. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ορισμένες σημαντικές προκλήσεις αφενός ε, την υποστήριξη μιας βιώσιμης οικονομίας που θα πρέπει να λάβει υπόψη να εγγυηθεί την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, την καινοτομία, την ενεργειακή επάρκεια, αλλά να δώσει και κοινωνικές απαντήσεις έτσι ώστε να απαντηθούν αυτές οι προκλήσεις σε σχέση με τα μεγάλα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε παγκόσμιο επίπεδο όπως οι κλιματικές αλλαγές, η ε, ανεργία, η κοινωνική ενσωμάτωση για να δώσουμε απάντηση στις γενικότερες προκλήσεις. Γιατί θα πρέπει να διατηρήσουμε θέσεις εργασίας, αλλά να δημιουργήσουμε και άλλες. Να προωθήσουμε λοιπόν την ενεργειακή αποδοτικότητα και γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις βιομηχανίες μας, τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες. καθώς και ορισμένες βιομηχανίες που έχουν περιφερειακή, περιφερειακό και τοπικό αντίκτυπο. Άρα, πιστεύω ότι αυτή η εξισορρόπηση μεταξύ καινοτομίας και διατήρησης βιομηχανιών ε, πρέπει να τύχει μίας αντιστάθμισης. Νομίζω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και στο τομέα, στον ενεργειακό τομέα, όπου μπορούν να συνταχθούν και άλλες βιομηχανίες που αφορούν την βαριά βιομηχανία, τις μεταφορές, την θέρμανση, την ψήξη, την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και βιομηχανίες που σχετίζονται με το τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, τις νέες τεχνολογίες, την πληροφόρηση και την επικοινωνία και βεβαίως και εδώ εμπλέκονται και οι ανανεώσιμες πηγές. για να φτάσουμε σε καθαρές μορφές ενέργειας. Επιμένω όμως ότι έχουμε βιομηχανίες όπως τις ένδυσης, τις υπόδησης, κλωστοϊφαντουργικά, ε, καλωδιώσεις και ούτω καθεξής που έχουν ε, βαρύνουσα σημασία σε πολλές περιφέρειες των κρατών μελών μας όπου θα μπορούσαν να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας ιδιαίτερα για τις γυναίκες. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτές τις ε, ιδιάζουσες καταστάσεις, πώς δηλαδή να συμφιλιώσουμε την καινοτομία με τις ε, βιομηχανίδες που ήδη προϋπάρχουν, καθώς και τη δημιουργία νέων. Αυτές είναι ορισμένες προκλήσεις που θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη και θα ήθελα να ακούσω και τι έχουν να πούν οι συνάδελφοι και επίσης το θέμα των ΜΜΕ στον βιομηχανικό τομέα. Πώς θα μπορούσαν να τύχουν υποστήριξης στα πλαίσια των ε, καινοτομιών. Τη στιγμή που αντιμετωπίζουν ε, χρηματοδοτικές ε, δυσκολίες. Κοινοτική στήριξη δηλαδή. και πώς μπορούμε να ε, ελαφρύνουμε τον γραφειοκρατικό φόρτο. Γιατί πολλές φορές αντιμετωπίζουμε δυσκολίες ε, στο να υπάρχει αυτή η χρηματοδοτική βοήθεια. Άρα να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, κάτι το οποίο δεν είναι ε, εύκολο, αλλά αποτελεί βασική πρόκληση, δηλαδή να διατηρήσουμε τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας και να δημιουργήσουμε και νέες. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά θα μπορέσουν να ληφθούν υπόψη για να έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με αυτά τα ζητήματα βαρύνουσα σημασίας για να υποστηρίξουμε τις ΜΜΕ και να προωθήσουμε ακολουθήσουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Αύριο προβλέπεται μία ακρόαση για το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Θα πρέπει λοιπόν να συσχετίσουμε την καινοτομία για να απαντήσουμε και όλα αυτά τα επιμέρους ζητήματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν ε, σύντομοι και θα ήθελα να παρακαλέσω ε, και τους δύο άλλους ομιλητές να κάνουν ακριβώς το ίδιο. Συνάδελφος πάντα είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ. Η παρούσα συζήτηση για την πράσινη οικονομία ή για την ε, οικονομία χαμηλού, χαμηλής ε, χρήσης άνθρακα είναι ε, ύψης σημασία, αλλά δυστυχώς δεν χρησιμοποιούμε παρά εφημισμούς. Παρά την επίκριση της στρατηγικής Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 βλέπουμε ότι η θέση της Επιτροπής είναι διφορούμενη. Όπως ε, ως Επιτροπή Ήτρε θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποιοι είναι οι στενοποί που, της βιομηχανίας και πώς θα μπορούσε η βιομηχανία μας να σταθεί νικητής χρησιμοποιώντας και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας για την ευημερία του μέλλοντος. Γνωρίζουμε την ανάγκη ε, της ε, αντιμετώπισης των ορεικτών καυσίμων και θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε ή να χρησιμοποιήσουμε γιατί αυτές τις πηγές ενέργειας δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα ορεικτά καύσιμα ε, έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα από πλευράς Κίνας, όπου έχει υπάρξει μία αύξηση της τάξης του 300%. Στόχος δεν είναι μόνο να μειώσουμε αυτή την κατανάλωση, αλλά να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πηγές σε λογικά επίπεδα έτσι ώστε να υποστηρίξουμε τον τομέα αυτό της βιομηχανίας. Γι' αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε την καινοτομία και να χρησιμοποιήσουμε σωστά και να ανακυκλώσουμε τις πρώτες ύλες. Αυτό θα πρέπει να είναι πάγιος κανόνας. Θα πρέπει λοιπόν να πραγματώσουμε αυτούς τους στόχους και να προωθήσουμε την ενεργειακή επάρκεια μειώνοντας τη χρήση του άνθρακα και να δούμε πώς μπορούμε να προβούμε σε συγκεκριμένες στοχοθετήσεις ε, η ταχύτητα και η εμβέλεια είναι ύψης τη σημασία. Υπάρχουν 24 εκατομμύρια επιχειρήσεις και εξαιτία των κλιματικών αλλαγών δεν πρέπει, να, πρέπει να έχουμε ένα χρονικό ορίζοντα 20 με 30 ετών. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να, επέλθουν, ε, να επισυμβούν αυτές οι αλλαγές και αυτό σημαίνει μεγάλη ε, προσπάθεια και από το επιστημονικό μας προσωπικό. Θα πρέπει να πω ότι η παρούσα κατάσταση ε, δεν οδηγεί σε, πάντα σε αναδιάρθρωση, στις αναγκαίες αναδιαρθρώσεις. Θα πρέπει να δούμε πώς έχουν τα υπάρχοντα μέτρα, αλλά να προβλέψουμε και νέα μέτρα, δηλαδή να έχουμε ε, έναν οικολογικό φόρο και να συνδράμουν οι επιχειρήσεις που μπορούν. Χρειαζόμαστε τεχνολογικές πλατφόρμες και μείωση των επιπτώσεων επί του περιβάλλοντος για να μην αρχίσουμε με τα κτίρια που έχουν μεγάλες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θα ε, προβάλλω πολλές ε, τροπολογίες που να έχουν λιγότερους εφημισμούς, αλλά και να είναι ιδιαίτερα στοχοθετημένες από τη δική μου ομάδα. Νομίζω ότι οι σωστές επιλογές θα μας καταστήσουν τους πρώτους για να ε, αναδιαρθρώσουμε την οικονομία μας. Ζανού. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχουμε να κάνουμε με μια συγκεκριμένη πρόκληση στο πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες ε, στα παραγωγικά μας μέσα. Βλέπουμε ότι στις παραδοσιακές ενεργειακές επιχειρήσεις ε, έχουμε δύο ε, θέσεις απασχόλησης ανά ένα εκατομμύριο ευρώ τζίρου. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε και τον τομέα των συλλογικών μεταφορών. Να δημιουργήσουμε δηλαδή νέες θέσεις εργασίας σε αυτούς τους τομείς που είναι τομείς του μέλλοντος, που είναι ήδη εν λειτουργία και μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας σε σχέση με τις παλαιές ε, βιομηχανικές δραστηριότητες. Υπάρχει μεγάλο δυναμικό. Σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα στην Ευρώπη. Αντιμετωπίζουμε ένα διτό ζήτημα, δηλαδή έχουμε μετεγκατάσταση βιομηχανιών αφενός και υπάρχει και η πιθανότητα να μετεγκατασταθούν και οι βιομηχανίες νέων τεχνολογιών. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο, ένα συγκεκριμένο σταθερό επενδυτικό πλαίσιο, γιατί πολύ συχνά βλέπουμε στα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα στη Γαλλία, ένα νομικό και διοικητικό πλαίσιο που είναι ασταθές, ιδιαίτερα για τις ανανεώσιμες. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να πλαισιώσουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα σε 10-15 χρόνια. Δεύτερον, να βοηθήσουμε τις ΜΜΕ να αναγνωρίζουν καλύτερα αυτή την πλαισίωση και να δουν πώς θα ασχοληθούν με στοχοθετήσεις. Γιατί πολλές φορές έχουμε και υπεργολαβίες που θα μπορούσαν να αποφευχθούν, ιδιαίτερα στο τομέα των αυτοκινητοβιομηχανιών. Αυτό αφορά και τον τομέα της αιωλικής ενέργειας. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τις ΜΜΕ να μπορέσουν να αναγνωρίσουν καλύτερα τους ε, επενδυτικούς τομείς. Και το θέμα των μισθωτών θα πρέπει να μας απασχολήσει, διότι πολύ συχνά στα κράτη-μέλη βλέπουμε ότι οι μισθωτοί χάνουν μια θέση απασχόλησης στους παραδοσιακούς τομείς και αναμένουν από μας να ασχοληθούμε με αυτούς έτσι ώστε να μεταταχθούν σε άλλους τομείς θα πρέπει να προωθήσουμε τις ε, επιχειρήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, να κάνουν δηλαδή και τις ανάλογες επενδύσεις. Στο τομέα των δηληστηρίων, ας πούμε, ξέρουμε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν ε, δις ε, εκατομμυρίων κέρδη, αλλά δεν βοηθούν τους μισθωτούς που χάνουν θέσεις εργασίας αντιστοίχως. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ως εκ τούτου κλείνουμε με αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και θα ήθελα να ρωτήσω τους ε, διερμηνείς ε, κατά πόσο μπορούμε να ξεπεράσουμε το ωράριό μας. Ε, και φτάνουμε στο σημείο 15 ε, δίνω το λόγο στον κύριο Λάγκεν. Ε, πρόκειται για την έναρξη της συζήτησης που σημαίνει ότι δεν πρέπει σήμερα να τα εξετάσουμε όλα τα θέματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόκειται για τον κανονισμό ε, Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την χρήση των νέων ελαφρών οχημάτων στο πλαίσιο της νέας οδηγίας για το διοξείδιο του άνθρακα. Από τον Οκτώβριο του 2009 προέρχεται η πρόταση, ήδη δηλαδή είναι πέντε μηνών. Αρμόδια είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος αλλά επίσης και η Επιτροπή Βιομηχανίας. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ το θέμα είναι πολύ σημαντικό για μας διότι όσον αφορά τις ε, οικονομικές και πολιτικές του πτυχές θίγει την μεσαία τάξη. Αυτά τα μικρά οχήματα ε, χρησιμοποιούνται κυρίως ε, από μικρούς επιχειρηματίες, από βιοτέχνες και πολύ λιγότερο από μεγάλες επιχειρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν οι επιπτώσεις από οικονομικές οικονομική και βιομηχανική πλευρά είναι πολύ πιο σοβαρές από ότι στην σχετική ρύθμιση για τα ΙΟΤΑΧΗ. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχουμε για το 2009 παγκοσμίω έχουμε περίπου 9,4 εκατομμύρια ΙΟΤΑΧΗ που παρήχθησαν και 10,8 εκατομμύρια ε, οχήματα μεγάλα και μικρά επαγγελματικά με μια ε, σημαντική διαφορά. Όσον αφορά τα επαγγελματικά οχήματα η Κίνα ήδη κατέχει περίπου το 50% της ε, παγκόσμιας παραγωγής. Στα γιοταχή μόνο 17% είναι το ποσοστό της Κίνας. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ είναι ένα θέμα ε, που ξεπερνάει κατά πολύ την πραγματικότητα. Η Κομισιόν λοιπόν έκανε μία πρόταση που βασίζεται στην, στον Οκτώβρη του 2000 για πάνω από 10 χρόνια. Η στρατηγική ήταν πάντα η αυτοδέσμευση. Ε, αυτό όμως είδαμε στα ΙΟΤΑΧΗ ότι δεν αρκεί. Και ως εκ τούτου εμείς ε, θέσαμε ένα πολύ φιλόδοξο στόχο που δεν άρεσε σε όλους εδώ στο Κοινοβούλιο, ε, δηλαδή να είναι 95 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο μέχρι το 2020 και η Κομισιόν με βάση αυτή τη νομοθεσία η Κομισιόν για τα μικρά επαγγελματικά οχήματα κατέθεσε σχετικές προτάσεις. Τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα της κατηγορίας υπαριθμών 1 έχουν 3,5 το μέγιστο βάρος και κατηγοριοποιούνται σε τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη έχουμε κυρίως γιοταχή, περαιτέρω εξέλιξη και το τρίτο στάδιο είναι αυτόνομες μεταφορές. Η προτάση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επειδή δεν έχουμε χρόνο θα είμαι πάρα πολύ σύντομο, η Κομισιόν προτείνει στόχος να είναι 175 γραμμάρια με face-in διαδικασία από το 2014 τον Οκτώβριο μέχρι το 2016. Και εδώ το εξή ερώτημα. Τι θα κάνουμε, κατά πόσον αυτά θα γίνουν παράλληλα με την νομοθεσία για τα γεωταχή ή κατά πόσο χρειαζόμαστε ειδικέ ρυθμίσεις. Εγώ λοιπόν θέλω να προτείνω ότι όσον αφορά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου ίσως πρέπει να την επιμικρύνουμε. Μετά έρχεται ο μακροπρόθεσμος στόχος 135 γραμμάρια από το 2020 και εάν το συγκρίνουμε στα ΙΟΤΑΧΗ τα 120 γραμμάρια ήταν ο στόχος για την πρώτη φάση και τώρα έχουμε φτάσει στα 175 γραμμάρια. Στον μακροπρόθεσμο στόχο η Κομισιόν είναι πιο φιλόδοξη ε, και παίρνει τα 135 γραμμάρια αντί για το 150. Κατά πόσο μπορεί να τηρηθεί αυτός ο μακροπρόθεσμος στόχος αυτό είναι κάτι επί του πρέπει να συζητήσουμε. Κατόπιν έχουμε άλλο ένα ειδικό πρόβλημα, ε, τα οχήματα που παρασκευάζονται σε διάφορες φάσεις, όπου οι κατασκευαστές κατασκευάζουν μόνο ε, τον κινητήρα ε, και κατόπιν επανέρχονται άλλοι ειδικοί που προτείνουν μεμονωμένες λύσεις για το αμάξωμα και το κατεθείς εξής. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε. Η Κομισιόν πρότεινε μια προσωρινή λύση με βάση την οποία οι κατασκευαστές ε, θα πρέπει να αναλάβουν τη δέσμευση ε, περιορισμού των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα για το σύνολο του οχήματο. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε διεξοδικά. Ο τομέα τη αυτοκινητοβιομηχανία έχει πάρα πολλέ επιφυλάξει και προτείνει είτε να πάρουμε ένα μέσο όρο. Εδώ η Κομισιόν έδωσε δύο παραγγελίε για δύο μοντέλα, άρα δηλαδή και εδώ αναμένουμε τι λύσει τη Κομισιόν. Το επόμενο θέμα είναι τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα λοιπόν για τα οποία τσακωθήκαμε εμείς εδώ. Ε, τα πρόστιμα στα μικρά επαγγελματικά οχήματα είναι υψηλότερα από ό,τι στα γιοταχή. Τα πρόστιμα λοιπόν εφόσον ξεπεραστεί κάποιο όριο των γραμμαρίων θα είναι 120 ευρώ αναγραμμάριο. Σας λέω αυτό είναι υπερβολικό, το απορρίπτω γιατί κάτι τέτοιο θα κατέστρεφε ε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτά τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα θα τα καθιστούσε υπερβολικά ακριβά. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα κατά πόσον θα πρέπει να ε, χορηγούνται πριν ε, εδώ προτείνεται από την Κομισιόν μία διαβάθμιση που καλύπτεται από τη ρύθμιση για τα γιοταχή. Και το τελευταίο θέμα που θέλω να φέρω είναι εξαιρέσεις για παραγωγούς ε, μικρών οχημάτων εν σειρά. 22.000 αυτοκίνητα είναι ένας ενδεικτικός αριθμός. Το θέμα είναι κατά πόσο ο αριθμός αυτός ε, είναι αυθαίρετος αν υπάρχουν ποσοστά. Βέβαια δεν έχουμε τα επίκαιρα στοιχεία αλλά πάντως υπάρχουν κάποιες προτάσεις να σημειωθεί αύξηση. Να σας πω και κάτι από την πρώτη συζήτηση που είχαμε στις 17 Μαρτίου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Εκεί λοιπόν ο μακροπρόθεσμος στόχος αντιμετωπίστηκε επικριτικά η εναρμόνιση με τον κανονισμό των γεωταχή τέθη βέβαια επιτάφητος ε, και όσον ε, ε, συζητήθηκε επίσης το θέμα των πριμ και των δανείων η μεγαλύτερη αυστηρότητα στα 170, μέχρι τα 175 γραμμάρια αυτό προτάθηκε να προβλέπετε και κάποιο όριο ταχύτητος. Ε, αυτό προτείνεται και από την Κομισιόν να ενσωματωθούν ε, συσκευές ελέγχου και μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η πρόταση της Κομισιόν σε γενικές γραμμές ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση. Όμως σε μεμονωμένα θέματα πρέπει η πρόταση Κομισιόν να συμπληρωθεί και εμείς ε, πρέπει να προσπαθήσουμε εφόσον υπάρξει συμφωνία πρώτης ε, ανάγνωσης ε, να παραμείνουμε σε αυτή τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί για τα γιοταχή. Πρόεδρος, αγαπητοί συνάδελφοι, πέντε έχουν ζητήσει το λόγο αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτό θα το καταφέρουμε μόνο αν ο καθένας μιλήσει κατά το μέγιστο ένα με δύο λεπτά. Αλλιώς μετά οι διερμήσεις θα φύγουν. Ο κύριος Περίλο είναι ο πρώτος, ο οποίος είναι και σκιώδης εισηγητής. Αυτό που είπε ο Πρόεδρος το λαμβάνω σοβαρά υπόψη μου σχετικά με το χρόνο. Και θα ήθελα να πω μόνο λίγα λόγια ελπίζοντας ότι στις επόμενες συζητήσεις θα μπορέσουμε να εμβαθύνουμε σε αυτό το θέμα το οποίο κατά την άποψή μου όπως είπε και ο συγητής είναι πολύ μεγάλη σημασία. Θα ήθελα να πω ορισμένα θέματα που αφορούν ε, κυρίως ε, ε, στο μακροπρόθεσμο στόχο στα 135 γραμμάρια. Αυτό λοιπόν το όριο των 135 γραμμαρίων, ε, εφόσον επιτευχθεί, σίγουρα θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο εμπόριο και στην τεχνολογία που αυτή τη στιγμή ε, δεν γνωρίζουμε ακόμα τις πρακτικές εφαρμογές τους. Εξάλλου, υπάρχουν ε, και κάποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις αν λάβουμε υπόψη μας όλον τον κύκλο των εκπομπών. Ε, θα υπάρξουν και σημαντικές ε, επιπτώσεις όσον αφορά και άλλες παράγωγες δραστηριότητες. Κατόπιν τούτου, για μένα αυτή τη στιγμή δεν είναι λογικό να ορίσουμε ένα τόσο μακροπρόθεσμο στόχο χωρίς να έχουμε κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία, χωρίς να μπορούμε να αξιολογήσουμε ε, αυτό που ε, θα έπρεπε καταρχήν να κάνει η Κομισιόν. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η έλλειψη ασφάλειας που προκαλεί αβεβαιότητα και στην αγορά και στις επενδύσεις και θεωρώ ότι είναι απαραίτητο πριν ορίσουμε τόσο αυστηρά όρια να κάνουμε μια σοβαρή και ε, ουσιαστική αξιολόγηση και κατόπιν να ορίσουμε τους στόχους. Και κάτι άλλο που θέλω να πω σχετικά με τις επιφυλάξεις για το άρθρο 8 που προβλέπει τις ε, κυρώσεις ε, για υπερβολικές εκπομπές και για την ε, περίοδο από το 14 μέχρι το 18. Ας μην ξεχνάμε Είπαμε ε, ότι αυτό το πρόστιμο των 120 ε, ευρώ είναι υπερβολικό. Θα μπορούσαμε ανταυτού να έχουμε κατά νου ε, να επανέλθουμε στις, στα πρόσωπα που βλέπονται αυτή τη στιγμή για τα γετοχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, λέει ο Πρόεδρος. Η, η συγγήτρια έχει το λόγο, η κυρία Χόλε. Θα ήθελα καταρχήν να δεχτώ αυτά που είπε ο εισηγητής για τις ΜΜΕ. Παίρνουμε μεγάλη ευθύνη έναντι αυτών. Και για κάθε ευρώ που επενδύεται για τα μικρά φορτηγά, για τη μείωση των εκπομπών, θα υπάρξει ένα ευεργέτημα ευρώ για τον τελικό χρήστη και ίσως είναι ακόμα υψηλότερο το ποσοστό. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να μειώσουμε τις εκπομπές στα μικρά φορτηγά για να βοηθήσουμε τις ΜΜΕ που δίνουν μεγάλο αγώνα αυτή τη στιγμή. Αναμέναμε αυτή την πρόταση εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Το Φεβρουάριο του 2007 ήταν ένα από τα επιπρόσθετα μέτρα για τη στοχοθέτηση α, περνώντας από 120 στα 130 γραμμάρια για τα μικρά φορτηγά. Υπάρχουν πολλοί κατασκευαστές που έκαναν βελτιώσεις ε, ε, πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν και αυτό είναι πολύ θετικό σε σχέση με τα επαγγελματικά οχήματα Βεβαίως τα μικρά φορτηγά δεν είναι καταρχήν οχήματα. Δεν μπορούν να γίνουν αεροδυναμικά, έχουν ε, προαπαιτήσεις, υπάρχει και το θέμα φόρτωσης και ούτω καθεξής. Και όπως είπε ο εισηγητής, τα εμπορικά ε, οχήματα είναι διαφορετικά ως προς την κατασκευή τους, έχουν, ακολουθούν διαφορετικά στάδια κάτι το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Από την άλλη πλευρά, πολλές βελτιώσεις που έγιναν από το 2007 στις μηχανές diesel μπορούν να ισχύσουν και να μεταφερθούν στα μικρά φορτηγά. Τα τελευταία τρία χρόνια είχαμε ε, μία βελτίωση 20% ως προς τη μείωση εκπομπών από οχήματα diesel. Αυτό είναι πολύ θετικό σημάδι. Και ως προς τα ηλεκτρικά οχήματα, ακόμα και χωρίς αυτή την ομοθεσία, βλέπουμε ότι ε, κατασκευάζονται όλα ένα και περισσότερο, χρησιμοποιούνται και στη δική μου επικράτεια και επειδή ξέρω ότι μας πιέζει ο χρόνος, Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε 160 γραμμάρια μέχρι το 2016 και 125 γραμμάρια μέχρι το 2020. Κύριο Σταυνόσκη, και αυτός ε, είναι σκιώδης συγητής. Θα είμαι πολύ ε, σύντομος, ε, συμφωνώ με τον κύριο Λάγκεν, κυρίως στην αρχή που είπε ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί αν ορίσουμε πολύ ψηλέ ε, τιμές χωρίς να γνωρίζουμε τις ε, επιπτώσεις και για την ε, περαιτέρω συζήτηση. Νομίζω ότι ο συγητής πρέπει να έχει μεγαλύτερο περιθώριο να λάβει τα αναλυτικά δεδομένα που θα σημάνουν, θα σηματοδοτήσουν το τι ακριβώς θα προκύψει, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα αναλυτικά δεδομένα είναι πολύ σημαντικά και εμείς ε, δεν θέλουμε να προωθήσουμε μόνο τους δικούς μας στόχους. Εγώ θέλω να υποστηρίξω αυτά που είπε ο κύριος Λάγκεν. Ε, ευχαριστούμε πολύ, κύριο Ζαντό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με εκπλήσει διότι δεν φτάσαμε σε όλα τα συμπεράσματα στα οποία θα έπρεπε να είχαμε φτάσει ως προς τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Πρόκειται για ένα τομέα σε κρίση και σήμερα με συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών διαπραγματευόμαστε εξαιρέσεις σε σχέση με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, ιδιαίτερα με την Κορέα. Έχουμε να κάνουμε με έναν τομέα όπου ακριβώς επειδή θέλουμε να ικανοποιήσουμε τους κατασκευαστές ελαφρών οχημάτων, δεν διαθέτουμε μία βιομηχανία που να είναι καινοτόμος και ανταγωνιστική και δυνατή, που να παραμείνει στην Ευρώπη. Αυτό σχετίζεται με την προηγούμενη συζήτηση για τους τομείς που θα πρέπει να προωθήσουμε, αλλά είδαμε με την ενεργειακή και κοινωνική κρίση ότι οι κατασκευαστές πήγαιναν πολύ πιο μακριά σε σχέση με αυτό που είχαμε θέσει ως τους εκπομπές κανονιστικά, ενώ τώρα λέμε ότι οι κατασκευαστές δεν έχουν ε, φιλόδοξους στόχους, ε, δεν είναι ιδιαίτερα καινοτόμοι και ούτω καθεξής όμως στα ελαφρά οχήματα, είδαμε ότι οι κατασκευαστές ε, δεν αρκέστηκαν σε αυτούς τους στόχους από πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής πλευράς και γι' αυτό αντιμετωπίζουν και μεγάλη κρίση. Άρα τα 160 γραμμάρια και 120 το 2016 και το 2020 αντιστοίχως είναι στόχοι που είναι ρεαλιστικοί για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφος Μάκης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον προλαλήσαντα. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία και νομίζω ότι ο κανονισμός δεν είναι ούτε καν αρκούντος φιλόδοξος. Νομίζω θα πρέπει να έχουμε μια μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο για τα εμπορικά αυτά ελαφρά οχήματα. Θα πρέπει να προχωρήσουμε και να τα εξομοιώσουμε με τα επιβατικά οχήματα. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό καινοτομίας από πλευράς αυτοκινητοβιομηχανίας και νομίζω ότι δράσαμε κάπως αργά με αυτόν τον κανονισμό, διότι η Κίνα ε, προτρέχει σε σχέση με το μερίδιο της αγοράς που καταλαμβάνει και βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, πολύ μεγαλύτερες παραγγελίες από την Κίνα. Θα πρέπει λοιπόν να στραφούμε σε αυτό το τομέα και να επικεντρωθούμε στον τομέα των καινοτομιών που ήδη υπάρχουν στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Περισσότερη καινοτομία, πιο καθαρά οχήματα και να κρατήσουμε αυτούς τους φιλόδοξους στόχους. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μια εντελώς νέα βιομηχανία σε πολύ λίγα χρόνια. So, ich bedanke ε, κύριε Λάγκεν, θέλετε να ξαναμιλήσετε μισό λεπτό να έχετε καλοσύνη. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Εγώ θα καταθέσω την ε, έκθεσή μου στο τέλος της εβδομάδας και τότε θα μπορεί να μεταφραστεί. Σωστά αυτά που ελέγχθησαν ότι η πρόταση για τα γιοταχή προήγαγε τις ε, καινοτομίες γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει οι καινοτομίες να ληφθούν επαρκώς υπόψη ευχαριστούμε πολύ και τους διερμηνείς ε, που τους καθυστερήσαμε κατ' εξαίρεση Γεια σας, μέχρι θα τα πούμε αργότερα.